Κυρίες και κύριοι, bonjour. La Θα ξεκινήσω με κάποιες ανακοινώσεις. Η κυρία Καρολίν Νικάς μας ανακοίνωσε το τέλος της θητείας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθότι εξελέγει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Το σημειώνουμε και σύμφωνα με το άρθρο 7, παραγραφός 2, της πράξης όσον αφορά την ε, εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και το άρθρο 4, παράγραφος 4 ανακοινώνουμε ότι η θέση της είναι κενή από την 18 Μαΐου 2010. Από τις 12 Μαΐου ο κύριος Μακνίλαν Σκοτ ανήκει στην ομάδα των φιλελευθέρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε να περάσουμε αμέσως τώρα στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Θα ξεκινήσω αμέσως με την έκθεση Μαλκά. Πρόκειται για τον διορθωτικό προϋπολογισμό 01-2010 και κατόπιν έκθεση ΤΡΥΠΕΛ όσον αφορά τις προβλέψεις για τα έσοδα και τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2011. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Βλάντιμιρ Μάνκα για τέσσερα λεπτά.